Dear colleagues, I would like to start because our timetable is very tough in the afternoon. Please take a seat. Παρακαλώ καθίστε να αρχίσουμε. Πάρτε και τα ακουσιστικά σας να τα χρειάζεστε. Και τώρα θα μιλήσω γερμανικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε Ξεκινάμε την απογευματινή μας συνεδρία, μια κοινή συνεδρίαση με το εξωτερικών υποθέσεων. Ε, έχουν έρθει ορισμένοι από την Επιτροπή αυτή. Θα ήθελα να σας πω ότι η κυρία Κώστα ζητά συγγνώμη είναι μέλος της Επιτροπής ε, Πολιτισμού, αλλά δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ, γιατί δυστυχώς ε, οι εορτασμοί για την 60η επέτειο από, την, ε, από τις συνθήκες δεν έλαβαν υπόψη τους δυστυχώς την ημερομηνία των συνεδριάσεών μας. Και η κυρία Κώστα τέλος πάντων έπρεπε να πάει στη Ρώμη σήμερα αλλά ξέρω ότι μαζί με την Τζούλη Βότς προετοίμασε την ε, συνεδρίαση αυτή και η Τζούλη Βότς θα την εκπροσωπήσει. Ευχαριστούμε την Τζούλη γι' αυτό και ε, ο Έλμαρ Μπρόκ, ο δεύτερος ηγητής, και αυτός σας ζητάει να τον συγχωρέσετε, θα καθυστερήσει για ένα 15 λεπτό. Αλλά επειδή το πρόγραμμά μας είναι αρκετά φιλόδοξο, θα ξεκινήσουμε και θα έρθει εκείνος ε, μετά από ένα τέταρτο. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το σημείο παρθμών 1 της ημερήσιας διάταξη. Είναι η έγκριση της ημερήσιας ε, διάταξης. Tagesordnung so genehmigt. Äh, Chairs Προέδρου, το σημείο 2 της διάταξη Έχουμε μετάφραση γερμανικά, γαλλικά, ολλανδικά, ισπανικά, ελληνικά, τσεχικά, λιθωνικά, πολωνικά, βουλγαρικά και σλοβενικά. Και Επίσης η συνεδρίαση ηχογραφείται. Τώρα, μια παρελθόν 3. Έχουμε τα πρακτικά της τελευταίας μας συνεδρίασης της 9ης Ιανουαρίου του 2017, τα οποία έχουν εγκριθεί. Έχετε καθόλου αντιρρήσεις, όχι. Άρα λοιπόν εγκρίνονται τα πρακτικά. Και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Ο λόγος για την διοργάνωση μιας κοινή συνεδρίασης είναι η έκθεση πρωτοβουλίας για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις. Από την ΑΦΕΤ η συγητής είναι ο Έλμαρ Μπρόκ και από την δική μας επιτροπή η Σίλβια Κώστα. οι δύο εισηγητέ ε, είχαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, την παρουσίασαν μάλλον στις, 9 Ιανουαρίου, λέγοντας σε ποια κατεύθυνση θέλουν να κινηθεί η έκθεση ε, και συζητήθηκε και οι δύο εισηγητέ ε, διατύπωσαν τις ιδέες τους σε ένα πρώτο σχέδιο, το οποίο είναι σημαντικό γιατί η σημασία του πολιτισμού στις ε, διεθνείς σχέσεις ε, είναι καθοριστική και εξελίσσεται. Λοιπόν, πριν ε, δώσω το λόγο στους ηγητές, θα ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Φίστησεν εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ε, θέλει να σας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχέδιο αυτό έκθεσης. Ε, όπως είπατε, ο πολιτισμός είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα ε, στις διεθνείς ε, σχέσεις. Πιστεύουμε ότι είναι ένας νέος τρόπος να προσεγγίσουμε τις διπλωματικές σχέσεις, την πολιτισμική διπλωματία, γιατί σημαίνει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων και θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, εισηγητές. Θα αρχίσουμε με την κυρία Ward, η οποία θα μιλήσει εκ μέρου της κυρίας Κώστα, που δεν μπορεί να είναι εδώ, για πέντε λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Έξι χρόνια, 60 χρόνια μετά από τη συνθήκη της Ρώμης, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις σε σχέση με την ειρηνική συνύπαρξη στον κόσμο. Προκλήσεις όπως ε, κρίση ταυτότητας και αξιών. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι παγκόσμιος παίκτη και να αξίζει το Νομπέλ Ειρήνης, πρέπει να ξαναρχίσει την προσπάθεια, ε, όμως να βασιστεί στις ε, πολιτιστικές, στις ε, αξίες και να προσπαθήσει να καταπολεμήσει κάθε ε, εξτρεμισμό ε, και ρατσιστική άνοδο. Χωρί την προώθηση των πολιτιστικών δικαιωμάτων, την πρόσβαση στη γνώση και στον πολιτισμό, χωρί ε, την ελευθερία ε, πολιτιστική έκφραση και πολιτιστικό διάλογο, δεν μπορεί να αναπαραχθεί ο πολιτισμό και ε, στι συγκρούσει υπάρχει ριζοσπαστικοποίηση. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία αναβίωση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών στρατηγικών στο πλαίσιο των 10 βασικών πρώτων τη προτεραιοτήτων. Ε, όσον αφορά ειδικότερα τις ε, πολιτιστικές ε, και δημιουργικές βιομηχανίες, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και της έρευνας η πολιτιστική ε, διάσταση ε, στον ψηφιακό τομέα και η πολιτιστική κληρονομιά και μέσω του ότι θα είναι το 2018 το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς ε, θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική ευκαιρία για να θέσουμε σε εφαρμογή αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα. Υπάρχει γενική συνένεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διεθνή πολιτική και ότι διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο λόγω στις πολιτισμικές υποθέσεις. Ε, χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα ε, που έχουμε τη σημερινή ε, συνεδρίαση γιατί είχαμε ζητήσει ε, το 2011 μία έκθεση που, ε, θα, που είχε ως αποτέλεσμα την, προσπάθεια πολιτιστικής ατζέντα που έλαβε χώρα το 2013-2014 υπό τις Ιταλικές και Λουξεμβουργιανές Προεδρίες συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια ζητήθηκε ένα πολιτιστικό πλαίσιο για την πολιτιστική διπλωματία νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντική η συνεργασία συνεργασία με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών, τον κύριο Μπρόκ, γιατί νομίζω ότι πρέπει να ε, μπούμε σε μια νέα φάση των διεθνών ε, πολιτιστικών ε, σχέσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την κοινωνία των πολιτών, αλλά πρέπει όλοι και κυρίως οι διεθνείς οργανισμοί, όλοι οι μηχανισμοί και οι φορείς σε συνεργασία σε πολιτιστικά θέματα να αποκτήσουν μια διαφορετική προσέγγιση. Ένα βασικό στοιχείο της ανακοίνωσης είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε μια επισκόπηση όλων των μέσων, των πόρων, των δράσεων και των ε, ε, ε, προοπτικών. Δηλαδή θεωρείται ο πολιτισμός ένας κοινό παρονομαστής. Εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση της ανακοίνωσης που θέτει τις εξής προτεραιότητες. Πρώτον, υποστήριξη της, του πολιτισμού ως βασικό κινητήριο μοχλό της ε, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, επίσης, προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου για τις ειρηνικές σχέσεις εντός μιας κοινωνίας, κάτι που επίσης το είχαμε πει και στην έκθεση τη δική μας για το διαπολιτισμικό διάλογο και το ρόλο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς επίσης, παραμένουμε δεσμευμένοι για την την ε, αξιοποίηση ε, της πολιτιστικής κληρονομιάς ε, και για, την, για τον τουρισμό αλλά και για την ανάπτυξη της οικονομίας. Πολλές πολιτιστικές, πολλοί πολιτιστικοί κλάδοι παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των κοινωνιών και η ΕΙΕΔ και τα, οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών ε, και οι πολιτιστικές ε, αντιπροσωπείες των κρατών μελών στο εξωτερικό και η UNESCO πρέπει να συνεργαστούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ τους, εντοπισμό εργαλείων και μέσων ε, για την συλλογή πόρων, προγράμματα όπως το Horizon 2020 και το Erasmus Plus να χρησιμοποιηθούν ως πλατφόρμα ανταλλαγή ιδεών ανεξαρτήτως ε, προέλευσης και πεπιθήσεων των ανθρώπων. Η στρατηγική όμως έχει περιορισμένο αντίκτυπο αν δεν έχει ως αποτέλεσμα συγκεκριμένες δράσεις και αυτά αποτελέσματα ή αν αυτά τα αποτελέσματα ε, γίνουν αισθητά μόνο στο απότερο μέλλον. Οπότε τέσσερις, ε, οι, βασικοί πυλώνες ε, της έκθεσης ε, ε, θα είναι η καινοτομία, οι δημιουργικές βιομηχανίες. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η κυρία Κώστα είναι Ιταλίδα, όπως θα θυμάστε. Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω τώρα. Είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση της συνεργασίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες εταίρους, να συνεχίσει ο διαπολιτιστικός διάλογος και ο διάλογος μεταξύ των θρήσκειων, ώστε να υπάρχει ελευθερία έκφραση έκφραση, ε, αμοιβαία κατανόηση, πολιτιστική ε, ποικιλία. Ε, πρέπει να, δεχθού, να, σεβόμαστε την επικουρικότητα και την αναλογικότητα στον τομέα του πολιτισμού και θέλουμε και την ανάπτυξη μια αποτελεσματική ενωσιακή στρατηγική για τι πολιτιστικέ σχέσει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και ένα πρώτο βήμα. Ζητούμε επίση την ενίσχυση των πολιτιστικών δικαιωμάτων ω τμήμα των αναντήρητων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να θεωρείται επίσης ένας εγκάρσιος πυλώνας μαζί με τα κοινωνικά, με τις κοινωνικές και τις περιβαλλοντικές πτυχές. Υπάρχει ένα τμήμα που αφορά τη διακυβέρνηση και τα εργαλεία. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις που αναφέρονται εκεί. Και τέλος, θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία ε, για την προσέγγιση ανθρώπου προς άνθρωπο. Είναι σημαντικά τα διασυνοριακά προγράμματα που πρέπει να θεωρηθούν σημαντικοί παίκτες για την μελλοντική ε, προσέγγιση ε, διαπολιτιστικού διαλόγου. Χρειαζόμαστε χαρτογράφηση των τοπικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών για να βελτιώσουμε την τοπική πρόσβαση στη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και την αποτελεσματική ε, συμμετοχή τους. Ε, να βασιστούμε σε μέσα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας και να λάβουμε υπόψη και την ισότητα μεταξύ των φύλων. Η Σίλβια είναι βέβαιη ότι θα συνεργαστούμε όλοι και εγώ είμαι βέβαιη, γιατί αυτό κάνουμε εμεί εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού και αυτό κάνουμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω του και όλου του συζητητέ εκ των προτέρων για την συμμετοχή του. Η κρίση που αντιμετωπίζουμε ε, σημαίνει κίνδυνο και προκλήσει, αλλά και ευκαιρίε. Ε, χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τι ευκαιρίε και α αδράξουμε την ε, ευκαιρία μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα ο κύριος Μπρόκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αφού άκουσα την ε, παρουσίαση, είμαι πεπισμένο ότι πρόκειται για μια θαυμάσια έκθεση. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσα πράγματα είχαμε συμπεριλάβει στην έκθεση. Αλλά πράγματι θεωρώ και θα ήθελα να το τονίσω ότι συμφωνώ ότι η πολιτική του πολιτισμού και στο επίπεδο των εξωτερικών υποθέσεων έχει καθοριστική σημασία. Είναι σωστό το οποίο υπόθηκε ότι η κουλτούρα, ο πολιτισμός είναι, αποτελεί ένα συνδετικό στοιχείο και βοηθάει στην επίλυση των συγκρούσεων. Το να αυτή η προσέγγιση της ε, κουλτούρας ας σαν κάτι το συνδετικό και όχι το διαχωριστικό μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό σε, πολύ, σε πολλούς τομείς και αυτό σε αντιδιαστολή με τα όσα βιώνουμε να γίνονται στις εξωτερικές ε, σχέσεις. Όταν πηγαίνω ε, στο εξωτερικό διαβάζω πάντοτε την ιστορία και κατατοπίζομαι για τον πολιτισμό της χώρας, γιατί ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, στις σχέσεις τις εξωτερικές. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορία και την οτροπία μιας χώρας, γιατί αυτό είναι, πολύ, είναι στοιχεία πολύ καθοριστικά και για την εξωτερική πολιτική μιας χώρας και οι πραγματικότητες εντός μιας κοινωνίας αλλά και μεταξύ των ε, χωρών ε, ε, εξαρτώνται πάρα πολύ από, το πολιτιστικό, από την πολιτιστική προσέγγιση. Ε, έχει υποθεί ότι οι ευρωπαϊκές κουλτούρες ε, έχουν κοινά στοιχεία κατά 4 πέμπτα και το 1 πέμπτο είναι αυτό το οποίο διαχωρίζει. Αλλά βεβαίως το 1 πέμπτο είναι αυτό το οποίο οδηγεί ορισμένα έθνη να θέλουν να ε, καθυποτάξουν τα άλλα. Και αυτή η προσέγγιση είναι ακριβώς στις ρίζες των εθνικισμών, του Βίλντερς και λοιπόν. Ε, παίρνουν ένα στοιχείο για, επί το οποίο προσπαθούν να τεκμηριώσουν γιατί η Γαλλία ή κάποιο άλλο έθνος ε, υπερέχει των άλλων. Εκεί που μας ε, διαφοροποιεί η κουλτούρα, αυτό δεν δικαιολογεί καμία υπεροχή. Αλλά οι διαχωρισμοί ε, απαρτίζουν τον κοινό πλούτο και θα πρέπει να συνενώνονται. Και αν κανείς έχει ακριβώς αυτή την κατανόηση, την ε, ενότητα μέσα από τις διαφορές, αυτή είναι μια δυνατότητα να πλησιάσει κανείς τον άλλον και να απαλείψει τις εντάσεις. Και αυτό το οποίο προσπαθεί ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι θέματα τα οποία εκμεταλλεύεται για προεκλογικούς λόγους προσπαθώντας να διαφοροποιήσει την εθνική και τη θρησκευτική ταυτότητα της χώρας του. Και γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η συνετή προσέγγιση του πολιτισμού έτσι όπως την ανέπτυξε είναι σημαντική θεωρώ ότι είναι μια σημαντική βάση την οποία εάν μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε σωστά θα μπορέσει να, έχει, να είναι εξίσου αποτελεσματική όπως άλλα αργαλεία. Για παράδειγμα όταν κάνουμε κάποιες ανταλλαγές ε, φοιτητών, ε, ακαδημαϊκές ανταλλαγές κλπ. Αυτές έχουν μακροπρόθεσμες ε, επιπτώσεις στην οτροπία ανθρώπων που μπορούν να διατηρήσουν για πολλά χρόνια μετά ε, και μέχρι και καθορίζει και την ε, στάση του έναντι της οικονομίας. Εάν ε, για παράδειγμα μηχανικοί έρχονται σε εμά και εκπαιδεύονται από τον Ειρηνικό ωκεανό ε, μετά από 30 χρόνια όταν θέλουν να παραγγείλουν κάποια μηχανήματα τα παραγγέλνουν από τη χώρα στην οποία έκαναν τις σπουδέ τους και υπάρχουν πολλές αποδείξεις ε, γι' αυτό. Ε, η κουλτούρα δεν είναι απλώς κάτι το όμορφο δεν είναι μόνο τα θέατρα, αλλά έχει απτές πρακτικές συνέπειες. Και γι' αυτό θα πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε ούτως ώστε οι διάφοροι ενεχόμενοι φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσουν την κουλτούρα και να τη συμπεριλάβουν στη χάραξη της πολιτικής τους. Οι χώρες ε, μέλη έχουν τις αντιπροσωπείες τους ε, στις διάφορες χώρες και εκεί θα πρέπει να εκπροσωπείται ο πολιτισμός στις άλλες χώρες. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα, ιδιαίτερα για μικρές χώρες, το Institut Français ή το Ινστιτούτο Goethe κλπ. Ε, ε, μπορούν ε, να ε, σταθούν εύκολα, αλλά οι μικρές χώρες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και να τους δώσουμε τη δυνατότητα οικονομικά να, παρουσιασ... να επιτείνουν την παρουσία τους στις άλλες χώρες. Αυτό ενισχύει τις ίδιες της χώρας και ενισχύει και την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία προβάλλει συνειδητά τις διαφορές μεταξύ των χωρών και τις διαφορετικές πολιτιστικές πραγματικότητες. Γι' αυτό ε, συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Κώστα. Και πιστεύω ότι θα πρέπει πραγματικά να ληφθεί υπόψη αυτή η πολιτιστική πλευρά και να αναπτυχθεί μια διπλωματία του πολιτισμού. Δεν πρόκειται μόνο για κάτι το ευγενές, αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά ε, μπορεί να προβάλλει και τα συμφέροντα των χωρών, το συμφέρον μιας χώρας. <clears throat> Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, τους δύο εισηγητές ευχαριστώ για τα εξαιρετικά σας ε, σχόλια. Ευχαριστώ πολύ και από τη δική μου πλευρά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους Σκιώδης. Και αν συμφωνείτε και κατά τα... Ένα, ε, σε αντίθεση με τις συνήθειές μας, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Αγγεμινές Παμπά από, την, από το Άλντε, η οποία πρέπει να πάει σε μια άλλη ακρόαση. Ευχαριστώ την κυρία ε, Σίλβια Κώστα και τον κύριο Μπροκ και ευχαριστώ την κυρία Ward που ε, εκπροσώπησε την κυρία Κώστα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις διεθνείς σχέσεις ε, μέσω του πολιτισμού. Μιλάμε για τις εγγενείς αξίες του πολιτισμού και το γεγονός ότι δημιουργεί γέφυρες μεταξύ ανθρώπων. Αυτές είναι οι αρχές που διέπουν την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι η κοινή δράση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετίζεται με τα κράτη-μέλη και τις χώρες εταίρους για να περάσουμε σε μία παγκόσμια τάξη ε, να προωθήσουμε την ειρήνη, τις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι προτάσεις, τροπολογίες που θα υποβάλω εμβαθύνουν ορισμένα ζητήματα οι σχέσεις πολιτισμού θα πρέπει να δώσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ε, επιστήμη, στην επιστήμη. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να προσδοθούν περισσότεροι πόροι στην διπλωματία και στην επιστήμη. Αυτό θα μας ε, επιτρέψει να προωθήσουμε την ε, διεθνή επιστημονική κοινότητα, την εξωτερική μας πολιτική και την διεθνή συνεργασία γύρω από την επιστήμη για να βελτιώσουμε και τις σχέσεις με τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ρόλο των πολιτιστικών Ινστιτούτων που προανέφερε ο κύριος Μπροκ ε, μέσω του ΕΟΝΙΚ. Η ΕΟΝΙΚ θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο. Εάν λοιπόν τα διεθνή αυτά Ινστιτούτα έχουν μία συγκεκριμένη δράση στην ε, εθνι, στις εθνικές μας χώρες θα μπορέσουν να παίξουν πολύ θετικό ρόλο στο ευρωπαϊκό πολιτισμικό αφήγημα. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε αυτή την διάδραση των ε, πολιτιστικών ε, Ινστιτούτων και ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ρόλο των πολιτιστικών επιτετραμένων στις πρεσβείες. Επίσης θα πρέπει να μιλήσουμε για την εκπαίδευση και, και την θρησκεία. Θα πρέπει βεβαίως όλα αυτά να συνάδουν με την ε, ανεξιθρησκεία και την ελευθερία ε, έκφρασης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Στην αρχή ξέχασα να αναφέρω ότι η συγγήτρια έχει το λόγο για τρία λεπτά, αλλά ε, τηρήσατε ακριβώς αυτά τα τρία λεπτά. Τώρα από το ΕΛΚ, κύριο Σταγερζεύσκη. Bardzo mi się spodobała Τι έχει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μία εγκάρσια και οριζόντια ε, προοπτική. Θα αρχίσω με τη ε, δική μου εμπειρία. Εγώ Ε, όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, ε, δέχτηκα τον Γάλλο και τον Γερμανό πρέσβη. Ο Γερμανός πρέσβης μου είπε ότι δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι οι Γερμανοί αποτελούν ε, αναπόστατο τμήμα της Volkswagen για παράδειγμα, αλλά θα πρέπει να ενδιαφερθούμε και για τον ε, Γκέτε, για τον πολιτισμό της Γερμανίας. Το ίδιο αφορά και τη ε, Γαλλία. Δεν είναι η Citroën, η Peugeot και η Renault, αλλά είναι και ο πολιτισμός, είναι και ο Μολιέρος. Όπως είπε και ο Έλμαρ, ο πολιτισμός είναι ένα εργαλείο για να επιληθούν ζητήματα, αλλά μπορούν να δημιουργηθούν και θέματα, δηλαδή ο πολιτισμός ενώνει αλλά και διαιρεί. Θα πρέπει μέσω του πολιτισμού όμως ε, να ε, δημιουργήσουμε δεσμούς και σε σχέση με την εκπαίδευση. Όταν ε, μιλάμε για πολιτική του πολιτισμού, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και εγγραφές που δεν είναι θετικές. Ο ίδιος ο πολιτισμός αποτελεί προστιθέμενη αξία καταρχήν, από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει ο πολιτισμός που χρησιμοποιείται ως μέσο για να προωθήσει άλλες αξίες που δεν έχουν σχέση με τον πολιτισμό αλλά με τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα μιας χώρας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφέροντα στοιχεία που μας απασχολούν και εδώ. Αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για το ρόλο των ΜΜΕ και εδώ το λέω υπό την ευρεία έννοια. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το, τέλο, το τέλειο μέσο το οποίο προωθεί ή αναχαιτίζει τον πολιτισμό. Μπορεί να οδηγήσει στην αποδοχή του διαφορετικού. Κάτι το οποίο σχετίζεται και με την ανεξιθρησκεία και με την ανοχή του διαφορετικού. Θα πρέπει λοιπόν να συμπεριλάβουμε διάφορες τέτοιες δράσεις στο πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κριστέ από την ΑΦΕΤ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, ευχαριστώ τους ε, συγκητές για το έργο τους. Το σχέδιο θέτει τα ορθά ερωτήματα και μας δίνει κάποιες κατευθύνσεις ε, για την πολιτική που θέλουμε να χαράξουμε. Εξετάζοντας το έγγραφο και ακούγοντάς σας, μπορώ να διαπιστώσω πολλά κοινά στοιχεία σε, στα θέματα τα οποία πραγματεύεται. Είμαι σίγουρος ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να καταλήξει σε ένα στεναρό κείμενο. Εγώ δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα στο σχέδιο. Πιστεύω στην ε, βαρύτητα, στη σημασία αυτού του θέματος. Ένα ζήτημα προτεραιότητας είναι αυτό των εργαλείων. Πιστεύω ότι το κείμενο είναι ξεκάθαρο όσον αφορά τους στόχους, αλλά είναι σημαντικό να οριστούν ξεκάθαρες ε, προτάσεις όσον αφορά την εκτελεστική πτυχή, ιδιαίτερα όσον αφορά ε, την πολιτιστική εκπροσώπηση. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι πόροι και πώς μπορούν να ενταχθούν οι προτεραιότητες αυτές ε, στον ε, προϋπολογισμό και στα εξωτερικά, και στα εξωτερικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Ένα άλλο θέμα αφορά τα περιβάλλοντα εντό των οποίων ε, κάποιες πολιτικές προσλαμβάνονται επιφυλακτικά λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης και εδώ θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη ενημερωτική εκστρατεία. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω αγαπητοί συνάδελφοι. Αναμένω με ανυπομονησία τη συνεργασία μας για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τζαμπάτσκι δεν βρίσκεται εδώ. Ο κύριος Τάνοκ από την ECR. Ούτε αυτός είναι εδώ. Από την ΚΟΕ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές για την προσπάθειά τους και θεωρώ ότι το σχέδιο καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό αρκετά από τα ζητήματα που απαιτούνται ώστε να αποκτήσει το πεδίο του πολιτισμού μια συνεκτική πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις. Από αυτή την άποψη συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας αναλυτικός απολογισμός των όσων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα στο πλαίσιο της Ατζέντα Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτισμό, ώστε να είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε παραπέρα τη στρατηγική μας. Να θεσπιστούν δηλαδή σαφείς και μετρήσιμοι κοινοί στόχοι και προτεραιότητες, αλλά και να αντιληφθούν διδάγματα από τις βέλτιστες πρακτικές. Οι στόχοι που απαριθμούνται στη στρατηγική είναι αρκετά φιλόδοξοι και απαιτούν τη συντονισμένη και την συνεκτική εργασία όλων των αρμόδιων φορέων. Αρχικά λοιπόν θα ήθελα να υπογραμμίσω το ρόλο που πρέπει να έχει ο πολιτισμός στην ανάπτυξη της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και γι' αυτό το σκοπό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση θα είναι επαρκής, με αυξητικό ρυθμό και θα αφορά κυρίως προγράμματα για την νεολαία. Από αυτή την άποψη συμφωνώ με την προτροπή του ψηφίσματος προς την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον πολιτισμό στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τη στήριξη των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ίση εκπροσώπηση μεταξύ των κρατών μελών και να καλύπτει το κενό που δημιουργείται σε χώρες όπως είναι η δική μου που βρίσκεται σε μνημόνιο και οι πόροι στον τομέα του πολιτισμού έχουν, ε, όπως είναι φυσικό, μειωθεί κατακόρυφα. Επιπλέον, ο πυλώνα του πολιτισμού θα πρέπει να προσθεθεί σε όλε τι υφιστάμενε και τι μελλοντικέ διμερεί και πολυμερεί συμφωνίε συνεργασία και να εξασφαλιστούν επαρκή πόροι και στελέχος των αρμόδιων φορέων και αντιπροσωπιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των στόχων. Πιστεύω επίση ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέρημνα στη διάσταση του πολιτιστικού τουρισμού η Επιτροπή θα μπορούσε να σχεδιάσει ένα ειδικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέσει πόρους αλλά και διευκολύνσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ενίσχυση της κινητικότητας και των ανταλλαγών με πολίτες των τρίτων χωρών και δεύτερων και να αναπτύξει σε διεθνές επίπεδο βέλτιστα προγράμματα, όπως είναι αυτό των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενισχύοντας έτσι του δεσμούς ανάμεσα σε πόλεις και περιοχές. Τέλος και κλείνοντα. Πιστεύω ότι δεν αρκεί από μέρου μα να μιλάμε, κυρία Πρόεδρε, μόνο για τη διατήρηση πολιτιστική κληρονομιά και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου τη. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να σεβαστούν την πολιτιστική κληρονομιά του κάθε λαού και να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους πολιτιστικά κοιμήλια και μνημεία, το οποίο είναι παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και εδώ θα μου επιτρέψετε να φέρω σαν Ελληνίδα χαρακτηριστικά την ε, επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα που διεκδικούμε ω Έλληνε πολίτε. Εκ μέρου λοιπόν τη ΓΚΟΕ θα καταθέσω τροπολογίε προ την κατεύθυνση τη βελτίωση του κειμένου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Helga Truppel για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, δύο εισηγητές και θα ήθελα να ευχαριστώ αυτό που είπε η κυρία ε, Ward ότι είναι ο τέταρτος πυλώνας ε, ο πολιτισμός της αϊφόρου ανάπτυξης και πιστεύουμε ότι θέλουμε πραγματικά να υπάρχει, είναι ένα σημαντικό τμήμα των διεθνών σχέσεων. Συμφωνώ και με αυτά που είπε ότι ο κύριος Μπρόκ ότι πρέπει να είναι μια ήπιας μορφής δύναμη ο πολιτισμός η ιδέα του πολιτισμού ποια είναι, γιατί ο Πολωνός συνάδελφος είπε κάτι σωστό, λέει ότι ο πολιτισμός μπορεί να συγκεντρώσει τους ανθρώπους αλλά μπορεί και να τους ε, χωρίσει. Οπότε καλό είναι να υπάρχει μια βασική κατανόηση του πολιτισμού και χρειάζεται μια ανοιχτή ε, δημοκρατική κοινωνία και όχι μια κοινωνία όπου κάποιοι αισθάνονται ότι είναι ανώτεροι από άλλους. Και αυτό το έχουμε δει και στο παρελθόν που έχει καταλήξει. Ε, είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι ε, να μπορούν σε δημοκρατικό επίπεδο να συνεργαστούν για τον πολιτισμό. Κάτι ακόμη, η κοινή προσέγγιση σε αυτή την ανακοίνωση πρέπει να είναι ότι δεν θέλουμε να εξαγάγουμε ευρωπαϊκές ή εθνικές, ε, ευρωπαϊκό ή εθνικό πολιτισμό, αλλά θέλουμε επικοινωνία και συνεργασία επιτόπου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τονιστεί περισσότερο στο κείμενο ότι το θέμα δεν είναι η, πολιτιστική, η παραδοσιακή πολιτιστική δημοκρατία, ε, διπλωματία, συγγνώμη, αλλά οι πολιτιστικές σχέσεις, συνεργασία με τον κόσμο, να συμμετέχουμε ε, στην προσπάθεια να, ε, κοινωνικής ένταξης ε, νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Οι ΕΙΕΔ πολύ, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, οι αντιπροσωπείες επίσης πρέπει να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία γιατί μπορεί μερικές φορές να δημιουργηθεί μια παραδοσιακή πολιτιστική διπλωματία. Εμείς όμως δεν θέλουμε αυτήν. Θέλουμε την άλλη ε, προσέγγιση, πραγματικές πολιτιστικές σχέσεις επιτόπου και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το μέσο αυτό να μην γυρίσουμε πίσω στην παλαιότερη προσέγγιση. Ε, η οίκη ευρωπαϊκής Κληρονομιά. Καλή ιδέα είναι αυτό όμως, γιατί για μένα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ σαφές ποια είναι η ιδέα πίσω από αυτό και γι' αυτό θα ήθελα να επανέλθουμε, να το επεξεργαστούμε για να εξασφαλίσουμε ότι αφορά τη συνεργασία, τη συμμετοχή άλλων ε, ενδιαφερομένων φορέων και πολιτιστικών οργανώσεων επιτόπου, να μην πάμε πίσω σε αυτή την παραδοσιακή προσέγγιση που είχαμε στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, τώρα εκ μέρους των ε, Πρασίνων από την ΑΦΕΤ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα επίση ε, να ευχαριστήσω τους συγητές για το έργο τους. Είμαι πεπισμένος ότι αν ο πολιτισμός αποτελέσει, αν θέλουμε ο πολιτισμός να αποτελέσει κινητήρια δύναμη, ο μόνος που μπορεί να το κάνει είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βασίζεται ακριβώς στην ε, πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, στην πρόθεση και την προστασία αυτής της πολυμορφίας. Και ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι σωστό να επισημαίνουμε ότι οι πολιτιστικές διεθνείς σχέσεις είναι μια στρατηγική η οποία πραγματικά συνάδει με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και τον τρόπο να προβάλλουμε την παρουσία μας σε όλο τον κόσμο αλλά επίσης επειδή ο πολιτισμός προωθεί μια μορφή διπλωματίας, μια ήπια διπλωματία η οποία βασίζεται στο διάλογο και οποία προωθεί την ε, ε, αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών. Ο πολιτισμός είναι λοιπόν ένας τρόπος να προαγάγουμε τα, τις ευρωπαϊκές ιδέες και αξίες και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου έχει μια πραγματικά προστιθέμενη αξία όσον αφορά τις διεθνείς μας σχέσεις. Και πιστεύω πραγματικά ότι θα πρέπει ο πολιτισμός να αποτελέσει κινητήρια δύναμη της στρατηγική μας ε, σε σχέση για παράδειγμα με τις γειτονικέ χώρες ούτε ώστε να οικοδομήσουμε πιο στέρες γέφυρες. That, uh, Επίσης πιστεύω ότι η έκθεση θα πρέπει να φωτίζει περισσότερο τη σημασία της διαπροσωπικής επαφής. Γιατί όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτού του είδους οι προσωπικές επαφές είναι το καλύτερο όχημα προκειμένου να προωθήσουμε την κατανόηση μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών, νοοτροπιών και τρόπων ζωής. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες δράσεις, ούτως ώστε να ενισχύσουμε τις ε, διαπροσωπικές σχέσεις για να προαγάγουμε την κατανόηση μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών. Και τέλος υπάρχει το θέμα του πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε ε, πώς μπορούμε να προβάλλουμε ένα κοινό μήνυμα προς τον υπόλοιπο κόσμο γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο να προαγάγουμε τις ε, 28 διαφορετικές ε, αξίες των χωρών μελών, αλλά το πώς να προβάλλουμε ένα κοινό μήνυμα. Αλλά επειδή τελειώνει ο χρόνος μου, θα ήθελα να θυμίσω ότι δεν έχουμε ένα ευρωπαϊκό τηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο θα ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να προαγάγουμε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπίλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτιστική ποικιλομορφία ε, διευρύνει τις επιλογές, ε, εμπλουτίζει τις ανθρώπινες αξίες ε, και ενισχύει την βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων, των πολιτισμών και όλου του κόσμου. Δεν το είπα εγώ. Είναι το τρίτο, η τρίτη σχέση της πολιτιστικής σύμβασης της UNESCO. Γι' αυτό ακριβώς την παράγραφο 5, όπου αναφέρεται ότι στον πολιτισμό πρέπει να γίνονται σεβαστές η αναλογικότητα και η επικουρικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, κάποτε μα είχε υποθεί από έναν συνάδελφο ότι δεν υπήρχε ε, ένα ευρωπαϊκό πολιτισμό αλλά πολλοί ευρωπαϊκοί πολιτισμοί, ο Γαλλικό, ο Ιταλικό, ο Ισπανικό κλπ. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό ε, μας δημιουργεί το δικό μα πλούτο. Η παράγραφο 7 για την απαραίτητη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά ε, την διατήρηση τη πολιτιστική κληρονομία και τη καταπολέμησης ε, ε λαθρέας, ε, ε, της λαθρεμπορίας πολιτιστικών ε, έργων είναι κάτι που πρέπει να, να το ενισχύσουμε επίσης. Θυμόμαστε για παράδειγμα τον τεράστιο σεισμό στην Ιταλία ε, και τις ε, που κατέστρεψε πάρα πολλά, ε, πάρα πολλά πολιτιστικά έργα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να αυξηθεί η πολιτιστική διπλωματία με μεγαλύτερη πρηματοδότηση, να υπάρχει πολιτιστική διπλωματία. Είναι καλό αυτό όπως ακούγεται, όμως ε, πρέπει να αποτελέσει ένα προνόμιο των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να προσπαθεί να ενισχύει τη θέση των κρατών μελών της σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να προσπαθήσει να ενισχύσει τις πολιτιστικές και ιστορικές σχέσεις μεταξύ των κρατών της και αυτό ε, μπορεί να είναι είναι πολύ εποφελές και για τις τρίτες χώρε και αναφέρομαι κυρίως στη σχέση για παράδειγμα της Γαλλίας με τις ε, ε, γαλλόφωνε χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλες δύο παρεμβάσεις. Τρεις, λέει Πρόεδρος. Ο κύριος Μελαμό. Ευχαριστώ πολύ <laughs> κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κώστα και τον κύριο Μπροκ για την έκθεσή της. Ήδη είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τον Ιανουάριο σε μια πρώτη ανταλλαγή από απόψεων. Ε, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να αξιοποιηθεί η κουλτούρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αξιοποιηθεί υπό την θετική έννοια για τις εξωτερικές ε, σχέσεις. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό όχημα και εργαλείο για να αναζητήσουμε, όπως είπε η κυρία Τρίπελ και ο κύριος Μπρόκ, ρίζες και τον ε, διάλογο βεβαίως εντός της πολυμορφίας. Εγώ είμαι μεταξύ αυτών που πιστεύουν ότι ο Θερβάντες, ο Μοντένι, ο Γκέτε, ο Ντάντε και ο Σέξπιρ δεν εξηγούνται μόνο από τη βάση τη εθνικής τους διάσταση, αλλά είναι Ευρωπαίοι συγγραφεί και είναι δύσκολο να σκεφτεί μόνο κανείς την εθνική τους ε, φυσιογνωμία. Ε, όλοι έχουμε το παρελθόν της, ε, το ελληνορωμαϊκό παρελθόν που είναι κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά. Επιτρέψατε μου να αναφέρω ένα συγκεκριμένο σημείο της έκθεσης, την παράγραφο 26, ε, όπου αναφέρονται οι πολιτιστικοί οδοί υπάρχουν και ε, τρίτες χώρες και χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, η Κωνσταντινούπολη έχει υπάρξει ε, πολιτιστική πρωτεύουσα. Είναι δυνατόν λοιπόν να συμμετάσχουν και τρίτες χώρες σε αυτά τα πολιτιστικά προγράμματα, στις πολιτιστικές διαδρομές. Ε, επίσης οι υποψήφιες χώρες ε, συμμετέχουν ε, σε αυτές τις πολιτιστικές διαδρομές και θεωρώ ότι είναι σημαντικές ευκαιρίες. Για να δείξουμε ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία. Το 2018 θα είναι το έτος το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει όσον αφορά τη χρηματοδότηση αυτών των πολιτιστικών διαδρομών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος, ο Χουντής από την ε, Επιτροπή Πολιτισμού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, διάβασα την έκθεση, άκουσα και τη συζήτηση είναι ένα ευχολόγιο, λέει καλά πράγματα, αλλά η εντύπωση που μου έδωσε είναι ότι κινείται εκτός πραγματικότητας. Τι εννοώ με αυτό. Και πριν πω τις παρατηρήσεις θέλω να σας πω ότι έχω θητεύσει και υπουργό Εξωτερικών. Έχω επισκεφθεί χώρες με διαφορετικούς πολιτισμούς και έχω κάνει διπλωματικές επαφές με τους διπλωμάτες διαφόρων χωρών. Στον τομέα λοιπόν αυτό δεν είναι τόσο ιδηλιακά τα πράγματα. Επανέρχομαι στο θέμα. Σωστά λέμε να μπει ο πολιτισμός μέσα στις διπλωματικές διεθνείς σχέσεις. Θεωρεί όμως δεδομένο ότι αυτό το πλαίσιο της διπλωματίας και γέννη των διεθνών σχέσεων της Ευρώπης είναι το σωστό. Είναι χωρίς ανομήματα. Πράγματι, η Ευρώπη, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στη γειτονιά που ζω εγώ, από την Ελλάδα, αλλά και στην περιοχή, προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα. Πολλές αμφιβολίες. Επομένως και η χρήση του πολιτισμού με μια αντίληψη υπεροχής απριόρι του ευρωπαϊκού πολιτισμού έναντι των άλλων πολιτισμών θα καταλήξει ο πολιτισμός, η πολιτιστική κληρονομιά, οι παραδόσεις, οι επαφές, οι αξίες να είναι συγκρουσιακό ή στο τέλος όπως επιβάλλεσε σε κάποιον πολιτικά, στρατιωτικά, να του επιβάλλεσε και πολιτισμικά. Πολλές φορές, το ζήσαμε σε άλλες εποχές, ο πολιτισμός μπαίνει μπροστά για να μπορέσει να διεισδύσεις και να επηρεάσεις ή να εκμεταλλευτείς τρίτες χώρες. Τα παραδείγματα από το, παρελθόν, μισό λεπτό, τα παραδείγματα από το παρελθόν είναι χαρακτηριστικά και διαπερνούν το, την Ευρωπαϊ, τις ευρωπαϊκές σχέσεις. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα, η νίκη της Αμοθράκης, η Αφροδίτη της Μήλου, τα περισσότερα μουσεία των κεντρικών ευρωπαϊκών πρωτευουσών που κατα, θα υλοποιήσουν αυτή την πολιτική είναι γεμάτα από, τέτοιες, ε, από τέτοια στοιχεία. Αλλά επανέρχομαι και για να τελειώσω, γιατί η πρόεδρος ενδεχομένως να μου πετάξει και το σφυρί, Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές αξίες. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταλήγω λοιπόν. Δεν έχουμε καταλήξει ή τουλάχιστον δεν υπάρχει κοινή παραδοχή. Θυμίσω τις έρηδες που ε, ήγηρε το προήμιο του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Συντάγματος σχετικά με τις καταβολές ε, τότε και που καταλήξαμε. Επομένως θα έλεγα η έκθεση έπρεπε αν θέλει και είναι σωστό να μπει όλο αυτό το πράγμα μέσα στις σχέσεις να πάει πιο βαθιά και να κάνει πιο ουσιαστικές ε, παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώ θα πρέ... Ε, πρέπει να είμαι τόσο αυστηρή γιατί έχουμε ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα. Ε, πυκνό πρόγραμμα. Δεν μπορώ να κάνω εξαιρέσει. Η Julie Watts για δύο λεπτά το πολύ. Και όχι, Julie, όχι η κυρία Κώστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ε, όλα αυτά που ακούσαμε ως τώρα και οι διαφορετικές απόψεις που εκπροσωπήθηκαν εδώ. Θα ήθελα απλώ να σας υπενθυμίσω ότι ο πολιτισμός δεν είναι κάτι το ε, σταθερό ε, ο πολιτισμός σημαίνει ότι δημιουργούνται και νέα πράγματα ε, και πρέπει να εμπιστευόμαστε τους καλλιτέχνες και τις κοινότητες, τις πολιτιστικές, γιατί ε, αυτό το κάνουν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και θα ήταν πολύ χρήσιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθουσε να το παροτρύνει αυτό, να το ενθαρρύνει, ε, να το γνωρίζουν περισσότερο αυτά τα κράτη-μέλη. Οπότε οι νέες πολιτιστικές μορφές είναι αυτό για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω. Ο πολιτισμός μπορεί συχνά να είναι μια διαδικασία επούλωσης ε, ε, δεν έχει σημασία αν μιλάμε για στρατιώτες, για μετανάστες, για ανθρώπους ε, που δεν ε, μπορούν να επικοινωνήσουν στην ίδια γλώσσα. Ε, οι άνθρωποι που πηγαίνουν από χώρα σε χώρα, η θίαση για παράδειγμα, αυτό το κάνουν πάρα πολύ καλά και δίνουν την ψυχή τους σε αυτό. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς, όχι μόνο για να δούμε κτίρια και ωραίους χορούς και παραδόσεις, πρέπει να έχουμε τη γνώση ότι ζούμε σε μία ε, ε, ήπειρο στην οποία έχουν συμβεί τρομερά πράγματα και δεν πρέπει να ξανασυμβεί αυτό λόγω της αύξησης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, ε, του λαϊκισμού. Ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς να επιδημήσουμε στον κόσμο ότι ο πολιτισμός είναι μία δύναμη υπέρ του καλού. Μερικές φορές ε, μιλάμε για τον πολιτισμό ως ε, κάτι που επιλύει τις συγκρούσεις, για παράδειγμα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πολιτισμός μπορεί να παρεμποδίσει ε, τις συγκρούσεις. Όταν έγινε η πλημμύρα στη δική μου περιφέρεια το 2015, ε, δεν, είναι μια περιφέρεια ε, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερη ποικιλομορφία, όμως ήρθα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 ενώσει βοήθεια ε, μουσουλμάνος από το Μάντσεστερ και ήταν οι πρώτοι που ήρθαν, έφεραν μαζί τους τον πολιτισμό τους, το φαγητό τους, τη γενεοδορία τους ε, και εγώ ήμουν σε μια εκκλησία ε, εκεί ο, ο Μουλάς και ο ιερέας μαζί συνεργάστηκαν για να μπορέσουν να δώσουν φαγητό στον κόσμο. Θα, μπορούμε να το κάνουμε αυτό όταν τα πράγματα είναι καλά τότε μπορεί τα πράγματα να μην ε, γίνουν άσχημα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό μόνον. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ... να πω ότι συμφωνώ πολύ με τη Judy Ward είναι σημαντικό ότι ο πολιτισμός όχι μόνο βοηθάει στην επίλυση των ε, συγκρούσεων, αλλά βοηθάει στην κατάργηση των στερεοτύπων. Ε, θα πρέπει να διορθώσουμε την εικόνα που έχουμε για τον άλλον. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ακριβώς αυτές τις ε, διμερείς ε, συναντήσεις, τις πολιτιστικές διαργανώσεις, οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει τις ε, σχέσεις σε τοπικό επίπεδο. Και έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δώσει κονδύλια, να χρηματοδοτήσει διάφορα προγράμματα με αυτά τα χρήματα. Στην έκθεση δεν νομίζω ότι αναφέρεται η πολυγλωσία σαν πολιτιστική διάσταση και νομίζω ότι θα έπρεπε να προσθεθεί. Ευχαριστώ πολύ και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι η 29 Μαρτίου 12 το μεσημέρι. Ε, μια πρώτη συνάντηση των εισηγητών θα γίνει στις 27 Απριλίου στις 9 και ο έλεγχος των τροπολογιών, εκεί όπου όλοι μαζί και πάλι θα τη συζητήσουμε, θα γίνει στις 3 Μαΐου και στις 30 Μαΐου θα αποφασίσουμε για την έκθεση μια κοινή συνεδρίαση. Αυτό είναι κάτι καινούριο για την Επιτροπή Πολιτισμού, ενώ τα μέλη της ΑΦΕΤ το γνωρίζουν, ότι στην παρουσίαση της έκθεσης οι ε, καλούν κάποιους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι δίνουν τη δική τους άποψη για τις εκθέσεις και οι δύο εισηγητές κάλεσαν σήμερα εμπειρογνώμονες και θα ήθελα να καλασορίσω θερμά τον πρέσβη κύριο Νικολά Μπιντού από την πρεσβεία της Ελβετίας και την κυρία Μιχάηλοβιτς από την Ευρώπα Νάστρα, την κυρία Σουζάνε Χέν από το Ινστιτούτο Γκέτε και τον Στέφαν Γκίς, διευθυντή της... Όχι, λάθος λέει πρόεδρος. Ε, διευθυντής του οργανισμού τους ε, Ευρωπαϊκής ε, Ακαδημίας ε, Μουσικής. Ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθατε. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο και στη συνέχεια θα ακούσουμε τους συζητητές από την Οικονομική και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή καθώς και από την, ε, τις περιφέρειες. Οχτώ λεπτά έχει το λόγο πρέσβης. Αλλά αν γίνουν και δέκα δεν θα σας μαλώσω. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που καλέσατε και την Ελβετία. Ε, θα σας μιλήσω πάρα πολύ σύντομα για το δικό μου οργανισμό που διαδίδει πάρα πολύ πολιτισμό ε, στο εξωτερικό. Θα μιλήσω με τον πολιτισμό και θα πω μετά μερικά πράγματα επιπλέον. Η Ελβετία μέχρι το 2000 δεν είχε πραγματικά ανακοίνωση της πολιτιστικής διπλωματίας. Ε, χρειάστηκε μία κρίση για να πιεστούν το Κοινοβούλιο και η κυβέρνηση, να δημιουργηθεί μία εικόνα πολιτιστικής διπλωματίας ε, είναι στο Ομόσπονδο ε, Υπουργείο Εξωτερικών. Ε, όλες πρέπει όλες και τα 26 καντόνια της Ελβετίας πρέπει οπωσδήποτε να σέβονται αυτές τις αρχές. Έχουμε 45 άτομα στη Βέρνη, ερχόμαστε σε επαφή με, τους, με τις με τις πρεσβείες μας ε, έχουμε 230 προγράμματα σε 76 πρεσβείες το 2016 για την πολιτιστική διπλωματία. Επίσης ε, έχουμε και 120 κανάλια ε, κοινωνικών μέσων για να προωθήσουμε την εικόνα μας αυτή. Έχουμε επίσης και την ιδέα της, των οίκων της Ελβετίας. Βρίσκονται σε μεγάλες πλατφόρμες μέσων μαζικής ενημέρωσης για να διαδικαστούν διαδώσουν το μήνυμα σε σχέση με την Ελβετία. Το βλέπετε εδώ μπροστά σα. ο οίκο της Ελβετία στο Ρίο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του καλοκαιριού. Η ιδέα είναι η εξή. Η κυβέρνηση χτίζει αυτόν τον οίκο και το περιεχόμενο το προτείνουν τα 26 καντόνια και οι ελβετικές εταιρείε εντό των οποίων υπάρχει πολιτισμό, αθλητισμό, εκπαίδευση ε, και ε, πολιτική πάνω από χίλια άρθρα. Ε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διάδραση σε επίπεδο κοινωνικών μέσων και η ιδέα είναι η διάδοση ε, του πολιτισμού της Ελβετίας. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, ε, προσπαθούμε να διαδώσουμε την πολιτιστική μας εικόνα. Εδώ βλέπετε, για παράδειγμα, είναι ο Υπέρ Βεντρίν εκεί, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Εδώ δείχνει η στον κόσμο ότι η Ελβετία των ε, εικόνων ε, υφίσταται πράγματι. Ε, προσπαθούμε λοιπόν η Ελβετία να προωθηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Κάτι πολύ σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τις μελέτες της εικόνας μας βάσει της παρακολούθησης. Μία από τα, ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα που κάνουμε είναι το να επικοινωνεί κανείς το κενό, να μην ξέρουμε δηλαδή ποια είναι η εικόνα της Ελβετίας στις χώρες οποίες δραστηριοποιούμαστε. Εδώ βλέπετε για παράδειγμα την εικόνα της Ελβετίας το 2016 ε, έχετε για παράδειγμα τον τουρισμό, ε, την οικονομία, το, ε, ε, τους το, ε, ε, πολιτικά θέματα, τρόφιμα και βλέπετε και κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ εμφανές, είναι ο πολιτισμός. Το θέμα λοιπόν του πολιτισμού είναι ένα κενό μας, ένα μειονέκτημά μας, πώς λοιπόν μπορεί κανείς να βρει έναν τρόπο να μάθει περισσότερα από την Ελβετία, αν παράδειγμα θέλει να δουλέψει εκεί. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να επικοινωνήσουμε να δημιουργήσουμε μια θετική εικόνα της Ελβετίας για όλα τα ε, ε, θέματα που είναι σημαντικά για την εξωτερική πολιτική της Ελβετίας. Ε, προσπαθούμε όλοι όσοι με όσοι προσπαθούν να ε, ε, ε, κοινωνήσουν, να μεταδώσουν αυτήν την εικόνα της Ελβετίας, να γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση επιτόπου και να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και των φορέων αυτών. Εμείς έχουμε πάντοτε ένα μείγμα μεταξύ της θεώρησης της Ελβετίας μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, των στοιχείων που θέλουμε να γνωστοποιήσουμε και της εξωτερικής πολιτικής. Οι στόχοι ως προς το κοινό είναι τα μέσα ενημέρωσης και όσοι αποφασίζουν, ας πούμε, ε, υπάρχει ένα ε, υπάρχει μια προσπάθεια για παράδειγμα ε, ε, μέσα, μέχρι και στο μετρό να προσπαθήσουμε να βρούμε στοιχεία για όλα αυτά, αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι προσδοκίες όλων όσων συνεργάζονται με την Ελβετία ξέρουμε την Ελβετία των στερεότυπων αλλά θέλουμε για παράδειγμα να γνωστοποιήσουμε και άλλα πράγματα οι επιστήμες, η εκπαίδευση η κατάρτιση και ο πολιτισμός. Η Ελβετία δεν είναι τόσο πολύ γνωστή για αυτά τα πράγματα. Και για να ολοκληρώσω, ε, ποια είναι η κατάσταση της ε, ιδέας της ε, Ελβετίας στον τομέα του πολιτισμού. Έχουμε λίγο, λίγους καλλιτέχνες που μπορούν να ενσαρκώσουν την ελβετική κουλτούρα, όμως έχουμε μουσεία, έχουμε φεστιβάλ, έχουμε πολύ μεγάλη παράδοση στην αρχιτεκτονική και στο σχεδιασμό, έχουμε υπέρ και κατά, στο πλαίσιο αυτό Τη προσπάθειας, προσπαθούμε να αναπτύξουμε την πολιτιστική διπλωματία μας. 30% ε, των ατόμων γνωρίζουν ε, την προσπάθεια ε, αυτή. Εμεί δεν είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε τόσο, τη βοήθη, να βοηθήσουμε τόσο τα έργα των καλλιτεχνών. Θέλουμε κυρίως να τα μεταδώσουμε, να τα διαδώσουμε και αυτό είναι ένα, ένα αυτό εγγράφεται στο πλαίσιο τη δημόσια διπλωματία. Θέλουμε α πούμε στο πλαίσιο μιας μια συνάντηση ενό φεστιβάλ. Τα πάντα αυτά έχουν μια, έναν αντίκτυπο. Πώς μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε μια πλατφόρμα που υπάρχει και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο της. Ε, για μας ε, η ισχύς ε, ε, της ε, ε, επικοινωνίας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν το έχουμε αυτό, λίγοι καλλιτέχνες θα θελήσουν να συνεργαστούν μαζί μας. Δεν θέλουμε να καλύψουμε βέβαια τα πάντα. Έχουμε και το πρόβλημα των γλωσσών. Έχουμε τρεις γλώσσες στην Ελβετία. Προσπαθούμε λοιπόν με το οπτικουστικά μέσα να λειτουργήσουμε αφήνοντας κατά μέρος έτσι το πρόβλημα των γλωσσών ε, και η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα είναι κάτι το πολύ ε, σημαντικό, όμως έχει και τους περιορισμούς τις Μερικές φορές ε, δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας. Και κάτι τελευταίο οι διεθνείς σχέσεις είναι δύσκολο να τις κατανοήσει κανείς. Ε, ναι, πρέπει να επικοινωνούμε, ναι, πρέπει να είναι μια ήπια δύναμη. Σήμερα πρέπει να αναπτύξουμε μια έντονη δημόσια ε, διπλωματία. Αυτό που λέει η Ευρώπη μπορεί να το πει και η Ελβετία. Αυτό που είναι δύσκολο όμως και περίπλοκο είναι να μιλάμε για διάδοση του πολιτισμού, λίγο περισσότερο για διάδοση, γιατί αυτή θα σας δώσει τη δυνατότητα να ενθαρρύνετε την, ε, αυτό το soft power, την ήπια εξουσία ε, ε, πρέπει λοιπόν η πολιτιστική πτυχή με την πτυχή της επικοινωνίας να, να συνδυάζονται. Να ξέρουμε επίσης ποια είναι η ιδέα της, ε, ε, η, θεώρηση της ευρωπαϊκής κληρονομιάς σε όλο τον κόσμο. Είναι διαφορετικά δύνατον να έχουμε μία διεθνή, να έχουμε σωστή, σωστές, σωστές διεθνές σχέσεις από αυτήν την έννοια. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς γίνεται αισθητή η Ευρώπη, το people to people ε, είναι ε, ε, πολύ εύκολο αν γνωρίζουμε για ποιους δουλεύουμε. Εμείς είμαστε ένα μοσπιδιακό κράτος, 26 καντόνια. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Το κλειδί είναι μια κατάσταση επικερδής για όλους και τα 26 καντόνια πρέπει να αναγνωρίζουν, να αναγνωρίζουν την πλατφόρμα μας ένα ε, τη, σημασία του να υφίσταται και να πούν ναι θέλουμε και εμείς να συμμετέχουμε και εμείς πρέπει να δούμε ε, πώς θα το κάνουμε αυτό, πώς θα τα καταφέρουμε, πώς μπορεί ένα καντόνι ε, να ε, αναπτύξει το δικό του αφήγημα ε, να λέμε ότι ναι είμαστε αυτό το καντόνι αλλά είμαστε και ε, Ελβετοί ε, και μετά ανήκουμε και στην Ευρώπη. Νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε να το επιτύχουμε. Κάποιο μίλησε για τη σημασία της τηλεόραση. Πράγματι το Euronews θα έπρεπε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να είναι σύμμαχος σε αυτή της, επικοινωνία, επικοινωνίας γιατί θα σα βοηθούσε πάρα πολύ σε αυτά που θέλετε να επιτύχετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Χάλοβιτς για την Ευρώπα Νόστρα. Μιχαήλοβιτς, κυρία Μιχαήλοβιτς. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που καλέσατε την Ρόπα Νόστρα για να μιλήσει σε αυτή τη συνεδρίαση. Γνωρίζετε ότι είναι η φωνή της πολιτιστικής ε, κληρονομιάς ε, στην Ευρώπη. Ε, στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές ε, οργανώσεις ε, και πολλοί πολίτες που μεριμνούν για την πολιτιστική κληρονομιά και είμαι χαρούμενη που μπορώ να τους εκπροσωπήσω. Όταν διοργανώθηκε το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Φόρουμ είχαμε δύο θαυμάσια νέα ότι ο Επίτροπος είπε ότι θα υπάρξει ένα Ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς και η κυρία Μογκερίνη είπε ότι θα υπάρξει μια δήλωση για τη χάραξη κοινή ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα του πολιτισμού. Ε, όλα αυτά ενίσχυσαν ε, τις ελπίδες μας γιατί πολλοί πολίτες ε, πρόκειται για μια συγκυρία που τίθεται να αμφιβόλω η ευρωπαϊκή ιδέα και είναι πολύ σημαντικό η ηγεσία της Ευρώπης να πει ότι λησμόνησε κάτι και θα πρέπει να τοποθετήσει τον πολιτισμό στον πυρήνα, στην καρδιά της ε, πολιτικής ε, και των εξωτερικών σχέσεων. Η Ευρώπη Νόστρα Χαιρετίζει λοιπόν την ανακοίνωση της Επιτροπής και θα ήθελα να καλέσω όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα οποία παρευρίσκονται εδώ πιστεύω να συνεργαστούν όσο να δυνατόν πιο στενά γίνεται για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή γιατί εδώ θα πρέπει να αναπτυχθεί μια συγκεκριμένη δράση και να γίνει ε, με σθένος και αποφασιστικότητα αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποδυναμώσουμε την ε, αρμοδιότητα των χωρών ε, μελών. Αντιθέτως, και η Ευρώπα χαιρετίζει το γεγονός ότι η δήλωση αυτή αναγνωρίζει την πολιτιστική κληρονομιά σαν ένας από τους τρεις βασικούς ε, πυλώνες. Η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Στρατηγική είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των δύο άλλων αξώνων που αφορούν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη καθώς και την ειρήνευση στις εξωτερικές σχέσεις. Τώρα, συγκεκριμένα σχόλια ως προς το σχέδιο της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, συγχαρητήρια προς τους δύο εισηγητές, τον κύριο Μπρό και την κυρία Κώστα, γιατί είναι πραγματικά φιλόδοξη η έκθεση, η φιλόδοξη το σχέδιο της έκθεσης και η μια ολιστική προσέγγιση την οποία στηρίζουμε, γιατί βεβαίως ο στόχος αυτής της στρατηγικής εν το γενάστε, δεν είναι μόνο μία διαφήμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του πολιτισμού, αλλά η συμβολή προς μία σε μια ε, ειρήνευση ε, όλου του πλανήτη. Και ε, θα ήθελα να αναφερθώ στον υψηλό συμβολισμό ότι έχουμε τη συνεδρίαση αυτή, την ερωτάσουμε σήμερα που είναι και η φλιβερή επέτειος των τρομοκρατικών επιθέσεων. Έχουμε σταδιακά συμπεριλαμβάνεται ο πολιτισμός σε όλες τις ε, πολιτικές της Ένωσης ως mainstreaming. Και γιατί ο πολιτισμός δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τις πολιτιστικές σχέσεις, αλλά σαν εργαλείο για όλες τις δράσεις που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, τον τουρισμό, τη γεωργία, την έρευνα και βεβαίως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τον επόμενο χρόνο ε, θα ορτάσουμε την επέτειο της Παγκόσμιας Διακήρυξης Ανθρωπίνων ε, Δικαιωμάτων. Και εδώ βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα άλλα κράτη ε, έχει να πει κάποια πράγματα εν σχέση με την σπουδαιότητα των πολιτιστικών δικαιωμάτων. Σημαντικό είναι να μην δοθεί έμφαση στις ε, διμερείς ε, σχέσεις μεταξύ των χωρών μόνον, αλλά στην αξιοποίηση όλων των εργαλείων της ε, πολυμερούς διπλωματίας. Και ορισμένοι βουλευτές ήδη το προανέφεραν. Οι ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες θα πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο σε όλες τις τρίτες χώρες, μέσα των πολιτιστικών Ινστιτούτων, αλλά και στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά όργανα των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν περισσότερο την πολιτιστική διάσταση στο έργο τους. Και θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει σαν ένα σημαντικός συνήγορος ε, για την ε, βαρύτητα ε, του πολιτισμού στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, Βεβαίω θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ήδη υπάρχει μια έκθεση για την πολιτιστική κληρονομιά. Η πολιτιστική κληρονομιά μετρά για την Ευρώπη. Αυτή είναι η δική μας έκθεση που τονίζει πιστικά, προβάλλει πιστικά δεδομένα όσον αφορά την καθοριστική σημασία του πολιτισμού. Παρακαλώ να αξιοποιήσετε και εσείς αυτά τα επιχειρήματα στις, στο επίπεδο των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχουμε το Ευρωπαϊκό Βραβείο για την πολιτιστική κληρονομιά. Και πάλι είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορείτε και εσείς να χρησιμοποιήσετε για την προαγωγή των βέλτιστων πρακτικών. Αριστεία, η ποιότητα στον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά. Ε, Μετά τον χρυσού αιώνα των ε, διεθνών συμβάσεων που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά, σήμερα αντιμετωπίζουμε μια ύφεση όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των συμβάσεων σε όλα τα επίπεδα. Και γινόμαστε μάρτυρες της ε, φιλελεύθερης, της υπονόμευσης αυτών των πολιτιστικών αξιών, όχι μόνο εκτός των χωρών, αλλά και εντό τη Ευρώπη. Για παράδειγμα, στη την πρώην Ιουγκοσλαβία από την οποία εγώ προέρχομαι. Θα πρέπει λοιπόν να επισημάνουμε το σημαντικό ρόλο της Ευρώπης όσον αφορά την ε, οικοδόμηση, την αποκατάσταση μάλλον ε, της κατεστραμμένης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ευρώπη δεν καλείται μόνο να παράσει τα κονδύλια, αλλά θα πρέπει να λάβει και ένα ηγετικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της εμπειρίας που έχει συσσωρεύσει η Ευρώπη εδώ και πολλές δεκαετίες, ε, αν όχι αιώνες, όσον αφορά την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά η πολιτική κληρονομιά απειλείται και σε εποχές ειρήνης. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να επικεντρώνουμε μόνο σε περιπτώσεις όπου καταστρέφεται η πολιτική κληρονομιά στο πλαίσιο έναπλων σειράξεων. Αλλά υπάρχει και μία μη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία δεν σέβεται την πολιτική κληρονομιά και την αφήνει να καταστραφεί. Και θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει σαν ένας στεναρός υπέρμαχος της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όχι μόνο συνεργασία με την UNESCO, αλλά και άλλα θεσμικά όργανα. Ακόμα και η Παγκόσμια Τράπεζα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως υπέρμαχος της πολιτικής κληρονομιάς. Η Ευρωπαϊκή ε, το ευρωπαϊκό έτος, η ευρωπαϊκή εποχή της πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι μια σημαντική ευκαιρία και θα έπρεπε να επιζητήσουμε να δημιουργήσουμε μια γέφυρα μεταξύ του έτους ε, αυτού και των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων, ούτως ώστε να υπάρξει να τονιστεί και ο ρόλος της ε, κοινωνίας των πολιτών, να δοθεί έμφαση στην ε, ε, διπλωματική, στη διαπροσωπική διπλωματία πρόσωπο με πρόσωπο. Επίσης, η εκπαίδευση στην ιστορία, όχι μόνο εντός της Ευρώπης, αλλά και εκτός της Ευρώπης. Τέλος, ε, όλα αυτά είναι τμήμα μιας, ενός νέου αφηγήματος για την Ευρώπη, που θέτει την πολιτιστική κληρονομιά στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, ελπίζοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να έχει έναν ευθύνοντα ρόλο στην ε, κινητοποίηση της πολιτιστικής ε, δέσμευσης σε παγκόσμια κλίμακα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους να τηρήσουν το χρόνο, γιατί αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε. Το Γκέτε, το Goethe. Και από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους δύο συγητές και βεβαίως θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας να μιλήσω σε αυτό τον κύκλο ως εκπρόσωπος των πολιτιστικών Ινστιτούτων και συνεπώς της κοινωνίας των πολιτών αναφέροντας την δική μας προοπτική και συγκεκριμένα πρακτικά παραδείγματα. Είναι μεγάλη τιμή. Θα ήθελα να επεσέλθω σε πέντε σημεία, εν συντομία, ε, περιγράφεται το επόβαθρο το οποίο μας οδήγησε στην ε, παρουσίαση της κυρίας Μογκερίνη όσον αφορά ε, τα πεδία που ο πολιτισμός μπορεί να είναι αποτελεσματικός στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τον όρο πολιτιστική διπλωματία και να, θα ήθελα να αναπτύξω τις ε, δικές μας ε, σκέψεις και συστάσεις. Η πρόταση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονων προσπαθειών να αποδοθεί στον πολιτισμό μια ε, ε, σημαντική θέση. Δύο σημαντικά έγγραφα, καταρχήν το θεματολόγιο για τον πολιτισμό του 2007, αλλά κυρίως η προπαρασκευαστική δράση μεταξύ του 2012 και 2014 κατά εντολήν αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η προπαρασκευαστική δράση μας οδήγησε σε σημαντικές γνώσεις και διατύπωση συστάσεων και θα ήθελα να κατονομάσω τα σημαντικότερα στοιχεία. Οι πολιτιστικές σχέσεις με τις τρίτες χώρες θα πρέπει να γίνονται σε ισότιμο επίπεδο. Ε, δεν θα πρέπει να γίνεται πολιτιστική εξαγωγή, αλλά συμπαραγωγή και ανοιχτός διάλογος που δημιουργούν εμπιστοσύνη μέσω της δικτύωσης. Ε, να είναι κανείς ανοιχτός και να ακούει τις ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών και των δημιουργών. Είναι το κλειδί για την επιτυχία. Η κουλτούρα χρειάζεται ελεύθερο χώρο και αυτονομία. Και επίσης χρειαζόμαστε μια στρατηγική για τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις και ένα επίσης κατάλληλο επαρκή προϋπολογισμό. Τέλος, διατυπώνεται η σύσταση, η εφαρμογή να εμπίπτει στην αρμοδιότητα εκείνων που έχουν ενεργό ρόλο στο χώρο του πολιτισμού. Ο πολιτισμός δεν είναι είδος πολυτελείας. Ο πολιτισμός είναι το μέλλον ιδιαιτέρως σε μια συγκυρία κρίσης και απώλειας της εμπιστοσύνης όπου χρειαζόμαστε περισσότερη συναισθηματική νοημοσύνη. Εμείς οι διαμεσολαβητές του πολιτισμού και δημιουργοί του πολιτισμού είμαστε υπέρ της ε, προβολής και της περαιτέρω αξιοποίηση του πλούτου του πολιτισμού γιατί ο πολιτισμός όχι μόνο προωθεί τις διαπροσωπικές σχέσεις, την εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών και την την πολιτιστική πολυμορφία. Ο πολιτισμός ε, χρησιμεύει για την πρόληψη των συγκρίσεων και την, τη συμφιλίωση και την ειρήνευση. Προωθεί την οικονομική ανάκαμψη, οδηγεί στη δικτύωση διαφόρων φορέων και διαφελάτει το, την ηλική και άειλη κληρονομιά μας. Κατά την εκπόνηση των πολιτιστικών προγραμμάτων είναι σημαντική διαδικασία και στη συνέχεια ε, ε, μπορούν να προκέψουν ε, εκπλήξεις. Ο πολιτισμός χρειάζεται συνέχεια, χρειάζεται βιωσιμότητα, μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη και η αίσθηση της κοινότητας. Θα ήθελα από διάφορους τομείς, εν συντομία και από διάφορες ε, περιοχές του κόσμου να κατανομάσω ορισμένα προγράμματα. Καταρχήν την Αφρική. Θέμα δημιουργική οικονομία. Στην Αφρική ζουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι κάτω από κρέα διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Η μουσική έχει μια ιδιαίτερη θέση στην Αφρική και σήμερα δεν ε, αποτελεί μόνο ένα πολιτιστικό παράγοντα, αλλά παρέχει, διανοίγει επιχειρηματικές δυνατότητες και δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης. Αλλά στην Αφρική υπάρχουν ε, ισχνοί πόροι και ισχνά μέσα για την ε, διασυνοριακή δικτύωση ε, και ανταλλαγή πληροφοριών. Γι' αυτό χρειαζόμαστε άλλου εταίρου από την κοινωνία των πολιτών και ε, δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα η οποία προσφέρει παρέχει σε 18 χώρες της Αφρικής δωρεάν αξιόπιστες πληροφορίες για την μουσική δημιουργία στην Αφρικανική Ήπειρο. Δικτυώνει τους μουσικούς, ε, καταγράφει διαφορά, καταχωρεί διαφορά άρθρα για την ε, μουσική καθημερινότητα στην Αφρική και δημιουργεί μια γέφυρα και προς την Ευρώπη. Το επόμενο θέμα αφορά την εργασία με τους μετανάστες περιοχές κρίση στην Εκεί Ανατολή για παράδειγμα. Όλοι γνωρίζετε ότι οι Σύριοι δημιουργοί ε, χρειάζονται την υποστήριξή μας, ιδιαίτερα στην εξορία. Η πολύμορφη πολιτιστική παράγωγη ε, έχει ζημιωθεί πάρα πολύ από τον πόλεμο. Εμείς υποστηρίζουμε με, μια μικρή, με ένα μικρό ταμείο με υποτροφίες, σύρους καλλιτέχνες σε πέντε κατηγορίες. Κινηματογράφος, θέατρο και performance, οικαστικές τέχνες, μουσική και λογοτεχνία. Και με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή τη, την ε, πολιτική κληρονομιά της Συρίας και θα διευρύνουμε αυτό το ταμείο και στην Ευρώπη, αυτό το πολιτιστικό ίδρυμα, Ούτε ώστε οι Σύριαν θέλουν να παρουσιάσουν το πολιτιστικό τους έργο στην Ευρώπη να βοηθήσουν στην κατάργηση των στερεοτύπων και να εντατικοποιήσουν το διάλογο μεταξύ μεταναστών και κοινωνιών υποδοχής. Ας μείνουμε όμως στις περιοχές κρίσης. Όλοι θα γνωρίζετε ότι ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τα παιδιά των μεταναστών, γιατί δεν θέλουμε καμία χαμένη γενιά. Βεβαίως θα πρέπει στα στρατόπεδα των μεταναστών να υπάρξει μέρη για την καθημερινή τους επιβίωση, αλλά αυτό δεν επαρκεί. Θα πρέπει να δώσουμε στους νέους ανθρώπους ένα μέλλον, να τους δείξουμε ένα μέλλον. Θα πρέπει να δώσουμε ερεθίσματα για τη φαντασία τους. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε τους ώστε τα παιδιά αυτά να μπορούν να ονειρεύονται. Γι' αυτό διανέμουμε δωρεάν στις περιοχές κρίσης. Στην Τουρκία, για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες στην Ιορδανία και στη Συρία για παιδιά μεταξύ 4 και 12 ετών, ε, βιβλία με εικόνες, ε, κλασικά βιβλία κλπ. Και μόνο τον περασμένο μήνα ε, μπορέσαμε να φτάσουμε σε 9.000 ε, παιδιά σε στρατόπεδα και διάφορα κέντρα. Υπόθηκε ήδη, υπόθηκαν κάποια πράγματα η κληρονομιά. Για μας είναι σημαντικό ε, σημαντική και η άλλη κληρονομιά, για παράδειγμα στην Ασία, στο Μπαγκλαντές και στη Δυτική Βεγγάλη μία πρωτοβουλία δημιουργήθηκε ε, μετά τον, τη διέρεση στη Βεγγάλη το 57 τότε 8 ε, εκατομμύρια άνθρωποι χρειάστηκε να μεταναστεύσουν από δύο πλευρές των συνόρων και ε, αυτό δημιούργησε μέχρι σήμερα πικρία, μίσος και αρνητικά συναισθήματα και αναμνήσεις οι παππούδες και οι γιαγιάδες ε, μετέδωσαν ε, σε επόμενες γενιές αυτή την πικρία. Ένα πρόγραμμα μεταξύ Ντάκα και Καλκούτας ε, κάνει έρευνες στο πεδίο της προφορικής ιστορίας και δημιουργήθηκε μια θαυμάσια εξαιρετική πλατφόρμα η οποία συνηγορεί υπέρ των κοινών στοιχείων και φροντίζει η τρίτη γενιά να μπορέσει να επεξεργαστεί ε, όλα αυτά τα νοητικά συναισθήματα που της παραδόθηκαν. Ε, τα, τους τελευταίους μήνες είχαμε πολλές συζητήσεις για το θέμα της πολιτιστικής διπλωματίας ή των πολιτιστικών σχέσεων. Εγώ, εγώ πιστεύω ακριβώς όπως η, ε, εγώ πιστεύω θα έπρεπε να ενισχυθούν οι προσπάθειές μας εδώ και σε σχέση με την ε, προπαρασκευαστική δράση που σας ανέφερα. Η πολιτιστική διπλωματία ε, στρέφεται προς το ζήτημα της εξαγωγής του πολιτισμού. Ε, δημόσιοι φορείς θέλουν να, μέσω πολιτιστικών προγραμμάτων να φτιάξουν το προφίλ τους. Ε, εμείς ως πολιτιστικά Ινστιτούτα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ένα πολιτιστικό διάλογο και να προωθήσουμε την κοινή ε, ε, αποδοχή. Πρόκειται για μια μακρά διαδικασία, η οποία δημιουργεί όμως βιώσιμα αποτελέσματα. Η παράκλησή μας ε, προς εσάς από την πλευρά της κοινωνίας των πολιτών. Χρειαζόμαστε μια περαιτέρω διευκρίνηση του ρόλου των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων και της εφαρμογής της ε, παγκόσμιας ε, πολιτιστικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε ένα χάρτη με προτεραιότητες στις διάφορες περιοχές. Ε, χρειαζόμαστε επίσης ένα προϋπολογισμό. Και θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα πρέπει... Όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτιστικών ε, προγραμμάτων, να το αφήσουμε στους ε, διάφορους ε, φορείς, αλλά θα πρέπει να δώσουμε δυνατότητα συνεργασίας όλων των οργάνων των αντιπροσωπιών της νεολαίας, των ιδρυμάτων κλπ. κλπ. Και η τελευταία μου φράση είναι η εξής. Χρειαζόμαστε ένα τακτικό έλεγχο μέσω δικτών και αξιολογήσεων του κατά πόσο η εφαρμογή της στρατηγικής βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα έρθουμε στον τελευταίο εμπειρογνώμονα, τον Στέφαν Γκρίς. Παρακαλώ να τηρήσετε και εσείς τα λεπτά. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και όπως ε, ακούσατε μιλάμε για την Ευρωπαϊκή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Οδείων και ε, ακαδημιών μουσικής, καθώς και μουσικών σχολών. Ε, εκπροσωπώ 300 ε, μουσικές ακαδημίες που καλύπτουν όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την Ευρώπη γενικότερα, δηλαδή 90% των θεσμών που εμπλέκονται σε αυτό τον τομέα και εκτός της Ευρώπης. Είμαστε ένα παράδειγμα μιας οργάνωσης που συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο δίκτυο. Βλέπετε στη διαφάνεια ποιοι, ήταν οι στόχοι του AEC. Ονομάζομαι Στέφαν Γκής, είμαι ο εκτελεστικός διευθυντής αυτού του οργανισμού και εγώ ήμουν διευθυντής μιας μουσικής ακαδημίας στη Γερμανία, αρχικά για πολλά χρόνια. Πώς κατανοούμε εμείς ε, την ε, παιδεία αυτή και την απόστολή μας. Μιλάμε για τη στρατηγική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις εταιρικές σχέσεις που χτίζονται σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Και αυτό είναι και το σημείο ύψης της σημασίας. Επίσης, αυτή η έκθεση ασχολείται και με επιπρόσθετα θέματα δηλαδή ο πολιτισμός ε, ε, περιέχει εγγενείς αξίες. Αυτό που έχει σημασία είναι ο καθένας να έχει πρόσβαση στην ε, πολιτιστική εκπαίδευση και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βεβαίως θα πρέπει να προωθηθούν πολιτιστικές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και τις τρίτες χώρες μέσα στα πλαίσια μίας προσέγγισης από τα κάτω προς τα πάνω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Κώστα και Μπρόκ που ασχολήθηκαν με αυτό το έγγραφο, το κατάρτισαν, που είναι ένα πολύ καλό έγγραφο εργασίας. Μιλάμε για δράσεις λοιπόν που είναι ρεαλιστικές και αποτελεσματικές. Δεν ε, συμφωνώ με την εκτίμηση που έδωσε ένας ευρωβουλευτής ότι πρόκειται για μία μη ρεαλιστική εικόνα. Αυτό δεν νομίζω ότι ισχύει. Όσο περισσότερο αμφισβητούμε τις ε, αξίες μας, τότε εμείς ως φορείς θα πρέπει να ενισχύσουμε την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα και αυτό μπορούμε να το κάνουμε πολύ επιτυχώς. Τώρα, επανερχόμενο στο έγγραφο, ένα από τα σημεία που θα ήθελα να τονίσω αφορά την ε, πολιτισμική μας πολιτική όπως οριοθετείται στην ατζέντα. Με κοινέ δράσεις έτσι ώστε και οι πολίτες να ξέρουν γιατί ευεργετούνται, καθώς και οι πολίτες τρίτων χωρών να γνωρίσουν καλύτερα τις ευρωπαϊκές αξίες. Η AEC δέχεται την εγγενή αξία της ε, καλλιτεχνίας ε, και πιστεύω ότι ανακύπτουν νέες θέσεις εργασίας και σε αυτό το τομέα για να συμμετέχουν οι άνθρωποι στην ε, πολιτιστική ζωή και να πλουτίζει ο άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή. Η AEC χαίρεται διότι τονίζεται και ο ρόλος της πολιτισμικής εκπαίδευσης και υποστηρίζουμε και την ε, διεθνή ε, το διεθνές στοιχείο του Εράσμους μέσα στα πλαίσια του ορίζοντα 2020. Ε, τι μπορεί να αλλάξει η Μιλάμε για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και τον ε, διασυνοριακό διάλογο καθώς και τις ευρωπαϊκές αξίες. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ρόλο μοντέλο και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η ελευθερία του καλλιτεχνικού εκφράζεστε. Ε, αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο γιατί αυτή η εγγενής αξία έχει μεγάλη σημασία αλλά και γιατί υπάρχει και καλλιτεχνική ελευθερία. Μιλάμε λοιπόν ε, για τη δυνατότητα του ανθρώπου να μπορεί να εκφραστεί μέσω των τεχνών. Ως προς την πολιτισμική συμμετοχή και την πρόσβαση στο πολιτισμό κάθε ανθρώπου, αυτό είναι ένα θέμα που μας είχε ήδη απασχολήσει Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να τονίσω ότι κατά την άποψή μας ε, ότι η εκπαίδευση στα γερμανικά Bildung μπορεί να προωθήσει ε, την ε, προώθηση των καλλιτεχνικών τομέων. Βεβαίως η καλλιτεχνική συμμετοχή αφορά όλους Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι και οι εμπλεκόμενοι φορείς ε, θα πρέπει να θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι έχει μεγάλη σημασία η εφαρμογή της σωστής πολιτικής της ευρωπαϊκής κληρονομιάς έτσι ώστε να προωθήσουμε την ε, καλλιτεχνική και πολιτισμική συμμετοχή όλα μας τα μέλη α, ασχολούνται με ελέγχους στα ε, σχολεία, στα, στους προσφυγικούς καταβλισμούς και οπουδήποτε αλλού μπορεί να προωθηθεί η μουσική. Μιλάμε ε, λοιπόν και για μελλοντικές κοινοτικές δραστηριότητες και γνωρίζουμε ότι μπορούμε να αναλάβουμε κοινωνική ευθύνη ε, εάν κανείς ε, προσπαθήσει να βγει από τον κλειό στον οποίο βρίσκεται, δηλαδή να μεταδώσει τις καλλιτεχνικές αξίες στον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαστε πολύ ακριβείς ως προς το χρόνο. Θα αναζητήσω από τους εκπροσώπους της ε, Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπή στον κύριο Απόστολο Κώστα. Βρίσκεται εδώ? Όχι, αλλά έχουμε τον εισηγητή από την Επιτροπή Περιφερειών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε εισηγητές, κύριοι εισηγητές, ε, κύριοι ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πρόσκλησή σας και γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα να ε, πούμε ορισμένα ε, πράγματα ε, για να αναφερθούμε στις πτυχές της εγκεκριμένης ήδη γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών όσον αφορά τη στρατηγική για τις πολιτιστικές σχέσεις. Κατά τη γνώμη μου, τρία στοιχεία θεωρώ πάρα πολύ πολύ ε, σημαντικά ε, και στα οποία θα ήθελα να επικεντρωθώ. Πρώτον, όπως αναφέρεται ε, στο σχέδιο γνωμοδότησης, είναι η σημαντική συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός κατά τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδιασμού, και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ε, της νοσιακής πολιτικής ε, για τις ε, διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι πιο κοντά στην κοινωνία. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε καλύτερα και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις ανάγκες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ε, ε, ε, των, κατοίκων. Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με τους εταίρους μας στο πλαίσιο της κοινωνίας και σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε πιο στοχευμένα και αποτελεσματικά προγράμματα ουσιαστικά επιτυγχάνοντας συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Βάσει των ε, δεδομένων αυτών ε, νομίζουμε ότι οι διατάξεις ε, που αφορούν τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην προσπάθεια αυτή πρέπει να απλοποιηθούν, να γίνουν ταχύτερε οι διαδικασίε, η άμεση πρόσβαση των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο υπάρχον πλαίσιο ε, συνεργασία και στα χρηματοδοτικά μέσα ε, των ε, θεματικών ενωτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να εξασφαλίζονται όλα αυτά. Επίση, η πρότασή μα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει την, την Επιτροπή των Περιφερειών ε, στη φάση του σχεδιασμού της στρατηγικής ε, και οι τοπικές και περιφερειακές και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της στρατηγικής βέβαια σεβόμενη την αρχή της επικουρικότητας. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, το δεύτερο βασικό ε, στοιχείο που προκύπτει από την γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών είναι η ανάγκη μεγαλύτερης σύνδεσης ε, του πολιτισμού ε, με την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε και νωρίτερα αυτό. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε στο ότι η πολιτιστική επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τεράστια. Μπορούμε μάλιστα να θεωρήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία πολιτιστική υπερδύναμη. Όμως έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την πολιτιστική μας διπλωματία και τις πολιτιστικές μας σχέσεις ακόμη περισσότερο σε συνεργασία με άλλες χώρες, κάτι που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόλο της Ευρώπης ε, ως ε, ισχυρού ε, παγκόσμιου παίκτη. Και το τρίτο και τελευταίο σημείο στο οποίο θα αναφερθώ σήμερα είναι η βασική διάσταση του πολιτισμού όσον αφορά τα βασικά ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πολλές περιπτώσεις, δυστυχώς, έχουμε δει ότι ο πολιτισμός θεωρείται εσφαλμένα συμπληρωματική πολιτική πολιτική ή πολυτέλεια και αγνοούμε η πολιτιστική η πολιτική μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο και στην αντιμετώπιση δύσκολων οικονομικών περιόδων με την ανάπτυξη ε, πολιτιστικών ε, ε, και άλλων κλάδων όπως για παράδειγμα ο τουρισμός και επίσης μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό σημαντικό ρόλο στη συνεργασία με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες μέσω ε, της πολιτιστικής, ε, των πολιτιστικών επαφών. Αν υπάρχουν περισσότερα κίνητρα προς τους νέους και ειδικότερα ε, σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, και ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε, για να μπορούν να συνεργαστούν ε, και να συμμετέχουν στον πολιτισμό και από την άλλη να ε, έρθουν σε επαφή με τις, απα, με τις ε, απαρέγκλητες αρχές στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να πω ότι ο πολιτισμός είναι βεβαίως ένας τομέας στον οποίο συνδέει τα κράτη και τους πολίτες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στον, με τον υπόλοιπο, στον κόσμο. η πόλεις και οι περιφέρειες που βρίσκονται ακριβώς ε, ανάμεσα στο βορρά και στο νότο ε, βρίσκονται σε πολύ πλέον εκτική θέση, οπότε θα θέλαμε να καλέσουμε εσάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμείνετε για το σημαντικό αυτό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε, εδώ ήταν ο εισηγητής της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Ε, θα πάρετε κι εσείς το λόγο για τρία λεπτά. Και δυστυχώς έχουμε και άλλα σημεία της ημερήσιας ε, διάταξης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ξεκινήσατε με μια Ιταλή συγγήτρια. Θα ολοκληρώσετε με έναν Ιταλό μιλητή εδώ εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ε, εμείς ε, ξεκινήσαμε το έργο μας, θα οριστικοποιήσουμε την έκθεσή μας και θα εγκριθεί κατά ε, το μήνα Μάιο και στην Ολομέλεια θα πάει. συμφωνώ με τα βασικά σημεία που παρουσιάστηκαν από τους δύο συγκητές, τον κύριο Μπρό και την κυρία Κώστα. Ε, ήδη έχουμε συνεργαστεί και πραγματικά συμμετείχαν σε μια πολύ ζωντανή συζήτηση και ακρόαση που διοργανώσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, χαιρετίζουμε την ε, δήλωση της, ε, την Ευρωπαϊκή Δήλωση ότι ο πολιτισμός είναι ένας βασικός ε, πυλώνας σταθερότητας και ειρήνευσης. Ο πολιτισμός έχει τεράστια σημασία όσον αφορά την προώθηση του βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, την ειρήνευση, άρθρο 3 της Συνθήκης αλλά θα πρέπει να πάμε να... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάει ένα βήμα παραπάνω και θέλει να εγκρίνει μια στρατηγική και να εφαρμόσει ε, τη στρατηγική και ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα δράσης. Δεύτερον, πρέπει να τονίσουμε το σημαντικό ρόλο του πολιτισμού στις εξωτερικές ε, σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο σαν εργαλείο ε, ήπιας ε, ε, ισχύω, αλλά σαν εργαλείο ειρήνευσης Γι' αυτό θα πρέπει η πολιτιστική διάσταση να συμπεριληφθεί ξεκάθαρα σε όλες τις ε, διαπραγματεύσεις για νέες ε, συμφωνίες. Για παράδειγμα με τις χώρες ΑΚΕ. Πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός θα πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως ως ο τέταρτος πυλώνας της βιώσιμης ανάπτυξης Τέταρτον, η κοινωνία των πολιτών, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ε, κατέχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο πεδίο του πολιτισμού. Αλλά θα πρέπει να επενδύσουμε στην υποστήριξη της ανάπτυξης μιας κοινωνίας των πολιτών στο πολιτιστικό πεδίο. Γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή ε, απευθύνει έκκληση για τη δημιουργία ενός φόρουμ ευρωπαϊκού πολιτισμού, ούτως ώστε να μπορούν όλες αυτές οι δυνάμεις να συμμετάσχουν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Πέμπτον, έχει επιτακτική σημασία να παράσχεται το πλαίσιο και τα εργαλεία του ώστε να υπάρξει πλήρη εφαρμογή. Ε, συμπληρωματικοί νέοι πόροι έχουν εγκριθεί για το Εράσμους ορίζοντας 2020 κλπ. Και τελευταίο σημείο θεωρούμε ότι η επένδυση στον πολιτισμό θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει τεράστιο κεφάλαιο για να αντιδράσουμε στην αυξανόμενη ε, πύρια της προπαγάνδας και του αφηγήματος του τρόμου, του φόβου. Ε, δεν είναι μόνο τα πολιτιστικά δικαιώματα αλλά και η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης που θα πρέπει να ενισχυθεί σαν ε, μια σημαντική διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ και για την συντομία της παρουσίασης ε, και νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτησή μας αλλά δεν θα ήθελα να παραλείψω να ρωτήσω την Επιτροπή αν έχει παρατηρήσει. Das Προφανώς δεν ε, ισχύει. Τότε θα ήθελα να ζητήσω από τους συγητές να μας πούν. Κύριε Μπρόκ. Πρέπει να πείτε παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι επικεφαλή της, ε, πολιτιστικού τομέα στην Γενική Διεύθυνση. Θα ήθελα να πω πόσο εκτιμούμε την υποστήριξη που έρχεται από το Κοινοβούλιο και επίσης αναγνωρίζουμε τον προκαταγωνιστικό ρόλο που έχει το Κοινοβούλιο στην ε, προπαρασκευαστική δράση που είναι αναγκαία για την πρόθεση αυτών των στοιχείων. Ε, πιστεύω ότι το στοιχείο κλειδί είναι ότι υπάρχει ένα πολιτιστικό μονοπάτι για τη βελτίωση των διεθνών σχέσεων που οικοδομείται στη βάση της αναγνώρισης των πολιτιστικών αξιών, της συνεργασίας και της αμοιβαίας ε, κατανόησης. Ε, θα ήθελα να σας καθησυχάσω. Δεν πρόκειται να επανέλθουμε στον παλαιό δρόμο της πολιτιστικής ε, διπλωματίας. Εμείς θα βασίσουμε την προσέγγισή μας στις πολιτιστικές ε, σχέσεις κυρίως. Maybe my colleague. yes, very short. Uh, head of unit. Um, Εγώ είμαι επικεφαλής ε, του τμήματος που αφορά ε, στη Γενική Διεύθυνση ΕΦΚΟ. θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση, την εκτιμώ πολύ και βρίσκαμε, βρήκαμε πολλά σημαντικά σημεία στο σχέδιο έκθεσης, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να πούμε, και αυτό φάνηκε και σε πολλές παρεμβάσεις, ότι παράγραφος 28 που αναφέρει τις ευάλωτες κοινότητες, στις ε, εξόχως απόκεντρες ε, περιοχές. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση ακριβώς σε αυτά τα ευάλωτα κομμάτια του πληθυσμού και να τα προστατεύσουμε σε καταστάσεις, ε, σε συγκυρίες κρίσης, γιατί εδώ ο πολιτισμός μπορεί να αποβεί σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης των κοινοτήτων και ε, δημιουργώντας ε, γέφυρες και με την ε, πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε όλους τους εμπειρογνώμονες, την, τους εκπροσώπους της Επιτροπής Περιφερειών, του, επίσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε σήμερα. Ο Έλμαρ Μπρόκ δυστυχώ, έπρεπε να φύγει, γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω την Τζούλι Βότς ω ε, Σίλβια Κώστα. Θε να πάρει το λόγο? Uh, I think so. Η Σίλβια θα ήταν πολύ ευχαριστημένη με τις σημερινές συζητήσεις. ως προς τη γενικότερη συνεργασία των ομάδων και των επιτροπών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εργασία μας, γιατί είμαστε πραγματικά δεσμευμένοι να δράσουμε στον πολιτιστικό τομέα και να ρίξουμε τα στεγανά που υπάρχουν. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, δεν είναι λεπτομέρεια θα πρέπει να ενταχθεί στις γενικότερες πολιτικές μας. Θα ήταν λοιπόν ιδιαίτερα ευχαριστημένη και όπως ξέρετε είναι ιδιαίτερα γενναιόδορη ως προς τη συνεργασία της με τους διάφορους εισηγητές για να λάβει υπόψη όλες τις τροπολογίες. Χαίρομαι που είχαμε και τους εμπειρογνώμονες μεταξύ μας και ε, χαίρομαι ε, γιατί μπόρεσα να λάβω το λόγο και στον χώρο όπου, δρούν όπου δρά η οργάνωση για τις ε, μουσικές ακαδημίες. Και γνωρίζω ότι κάνουν πολύ σοβαρή εργασία και στον τομέα υποστήριξης των προσφύγων. Ευχαριστούμε πολύ θα κλείσω με ένα παράθεμα του πρώην ε, Προέδρου Ιωάννης Ράου. Ο πολιτισμός ε, δεν είναι η σαντιγή πάνω στο γλυκό, αλλά η μαγιά στη ζύμη. Θεωρώ ότι είναι πολύ εύστοχη η λύση αυτή όσον αφορά τον ευρωπαϊκό μας ε, πολιτισμό και την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Νομίζω ότι και εδώ η μαγιά στη ζήμη θα συνέβαλε πάρα πολύ στην επιτυχία του γλυκού. Ευχαριστούμε λοιπόν. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε έναν πολύ καλό κοινό δρόμο. Θα ήθελα να ευχηθώ καλές διαβουλεύσεις στους συζητητές και τους σκιώδεις, καλούς συμβιβασμούς και στις 3 Μαΐου θα συναντηθούμε για μια κοινή συνεδρίαση και τώρα λοιπόν θα ήθελα να πω ότι λύεται η κοινή συνεδρίαση με την ΑΦΕΤ. Η δική μας συνεδρίαση Επιτροπής Πολιτισμού θα ξεκινήσει αμέσως και θα έρθουμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, εάν δεν απατώμε. Εδώ πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ελεκτρονικών Επικοινωνιών. Και εδώ η Κομισιόν ε, παρουσίασε ένα πολύ ε, ε, περιστατωμένο πόνημα. Αρμόδια επιτροπή είναι, επί είναι έχει και ειδικέ αρμοδιότητες ΙΜΚΟ και εμεί, ω Επιτροπή Πολιτισμού κάνουμε μια γνωμοδότηση. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους όσους εγκαταλείπουν την αίθουσα να το κάνουν το ταχύτερο δυνατό και ή δυνατόν ε, ήσυχα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Συγκριτής, είναι ο συνάδελφος κ. Μαλτέζης, τον οποίο θα ήθελα να δώσω αμέσως το λόγο με την παράκληση να μην μιλήσει περισσότερο από πέντε λεπτά, γιατί έχουμε δύο σημεία στην ημερήσια διάταση πριν ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Παρακαλώ.